Λοιπόν, τώρα στην εκλογή αντιπροέδρου. Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 17 και 20 του κανονισμού μας έχω λάβει τις εξής υποψηφιότητες. Ο συνάδελφος κύριο Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο που δέχτηκε την υποψηφιότητά του και προτέθηκε επίσης και αυτή δέχτηκε η κυρία Άνελη Γέτεν Μέκη. Οι δύο υποψήφοι μου ανακοίνωσαν ότι όπως σας είπα προτάθηκαν και δέχθηκαν την υποψηφιότητα Και η εκλογή θα γίνει με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να εξοικειωθείτε λιγάκι ε, με το ηλεκτρονικό σύστημα θα κάνουμε μια δοκιμαστική εκλογή. Όταν θα ξεκινήσει η ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι, η οθόνη θα δείχνει το τι ψηφίζουμε. Δηλαδή ε, θα ψηφίζουμε για τον υποψήφιο, ε, τον κατάλογο των υποψηφίων ε, και εσείς θα πρέπει να πείτε ποιον προτιμάτε πατώντας ε, το μπλε κουμπί και μπορείτε το κουμπί να το πάτε προς τα πάνω προς τα κάτω είναι ο cursor και εάν θέλετε ή βρήκατε τον υποψήφιο που επιθυμείτε εκεί θα πατήσετε το συν Αυτό το ρώτησαν πάρα πολύ. Αν θέλετε να δηλώσετε αποχή, διότι έχουμε δύο υποψηφίους, να πατήσετε το κουμπί που λέει αποχή. Είναι το μεσαίο κουμπί. Και στην περίπτωση αυτή, ναι μεν θα ανάψει το μπλε λαμπάκι, αλλά παρόλα αυτά εσείς θα έχετε συμμετάσχει στην ψηφοφορία δηλώνοντας αποχή. Είναι δυνατό να γίνει αυτό. Και βεβαίως μπορεί να μην θέλετε να συμμετέχετε στην ψηφοφορία. Αυτό είναι δική σας απόφαση. Προς ε, μεγάλη σας έκπληξη θα προτείνουμε για άλλη φορά δοκιμαστικά την Μονσέρα Καμπαγέ και η Γιουμίλια Τζόνσον. Αυτοί οι δύο ε, υποψήφια έτσι ενδεικτικά για να κάνουμε τη δοκιμή προφανώς. Ξεκινάμε λοιπόν με τη δοκιμαστική ψηφορία. Ψηφίστε, ψηφίστε τι θέλετε από τις δύο που σας ανέφερα. Βλέπετε λοιπόν στην οθόνη σας εμφανίζεται ε, election test. Θα ψηφίστε είτε την κυρία Μονσερά Καμπαγέ είτε την κυρία Μικέλε Τζόνσον. Μπορείτε να κουνήσετε τον κέρσορα προς τα πάνω ή προς τα κάτω και όσοι από όποιον θέλετε, όποιον προτιμάτε, θα κουνήσετε τον κέρσορα και αφού το βρείτε το όνομα και είναι κόκκινο, εκεί θα πατήσετε. Λοιπόν, ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Δοκιμαστικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι.

Ε, Κύριε Λούκα, θέλετε κι εσείς να δηλώσετε υποψηφιότητα. Παρακαλώ. Όχι, εγώ δεν θέλω να θέσω υποψηφιότητα, αλλά θα ήθελα οι δύο υποψήφοι να ε, συστηθούν λιγάκι, γιατί εγώ τη δεύτερη υποψήφια ούτε που την ξέρω. Κοιτάξτε κύριε Λούκα, δυστυχώς αυτό δεν προβλέπεται στο καταστατικό μας. Οι εκλογές γίνονται χωρίς ε, σύσταση των υποψηφίων. Πάντως ε, έλαβε υπόψη με αυτό που είπατε. Εν πάση περιπτώσει τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, τώρα θα βγουν τα ονόματα. Σπανό. Mm-hmm. So. Λοιπόν, βλέπετε τα ονόματα, έτσι δεν είναι, Καστάλντο και Γετενμάκη. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Ich frage, ob alle Ψηφίσατε, ψηφίσατε όλοι ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές. Ξαναρωτάω, ψηφίσατε όλοι για να κλείσουμε την ψηφοφορία, γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα ψηφίσατε, έτσι δεν είναι. Δεν κατάφερα να έχω αποτέλεσμα στο μηχάνημό μου. Δηλαδή. Τι εννοείται, δηλαδή εννοείται ότι δεν λειτουργεί η συσκευή σας. Dann warten wir τότε να περιμένουμε, να περιμένουμε να φτιάξουν τη συσκευή σας. Κυρία συνάδελφοι, πηγαίνετε στη θέση 253. Πάρτε την καρτέλα σας, πηγαίνετε εκεί στη 253 που είναι άδεια και ψηφίστε που είναι έτσι κι ε, και θέση των πρασίνων που δεν χρειάζεται να πάτε στο εξωτερικό. Αν θέλετε και το ΕΛΚΑ έχει να σας προσφέρει θέσεις, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είχαμε και ειδικού εδώ τη τεχνολογία που βοηθήσαν. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, τώρα ψηφίσατε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. 301 για την κυρία Γιατεμάκη, για τον κύριο Καστάλτο 285, άρα δηλαδή η κυρία Γιατιμέκη εκλέγεται. Ich Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τη συνάδελφο, αλλά δυστυχώ δεν με ακούει. Από ό,τι φαίνεται ούτε να τη συγχαρεί κανεί δεν μπορεί. Κυρία συνάδελφε, ε, σας συγχαίρουμε και σας καλωσορίζουμε στο Προεδρείο. Προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία. Κυρίε και κύριοι, όσον αφορά την ε, πρόταση τη διάσκεψη των Προέδρων για τι Ολομέλειε του 2016 που κοινοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό, δεν κατατέθηκαν ε, τροπολογίε. Γι' αυτό λοιπόν το ε, ημερολόγιο των Ολομελιών του 2016 εγκρίνεται. Το χρονοδιάγραμμα των Ολομελιών. Ζητώ συγγνώμη που έχω κρυώσει. Περνάμε τώρα στι ε, ψηφοφορίε. Αλλά αν έχει την καλοσύνη, λίγη υπομονή για να ε, συντονίσουμε λιγάκι το σύστημα των ε, ψηφοφοριών. Και ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες με την έκθεση STIR. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία. Συμφωνεί για το εμπόριο, την ανάπτυξη και την συνεργασία με την Νότια Αφρική. Έκθεση ΣΤΙΡ, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 623 υπέρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον κύριο Στύρ. Επόμενη έκθεση της κυρίας Σαρτζεντίνη και του κυρίου Κάρινης πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν ε, λάβαμε εδώ ε, πρόταση τροπολογιών. Κατόπιν τούτου εγκρίνεται και η θέση του Συμβουλίου, γιατί ούτε και από αυτής υπήρξαν τροπολογίες. Πάμε στην έκθεση Kirchhoff Simon. Ε, πληροφορίες που συνοδεύουν τις ε, μεταφορές χρηματικών ποσών. Και από αυτής της έκθεσης δεν λάβαμε τροπολογίες, ούτε προτάσεις για να απορριφθεί η θέση του Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου η έκθεση αυτή εγκρίνεται. Πάμε στην έκθεση Τσβέφκα, ε, διαδικασίες αφαιρεγγιότητας. Και εδώ δεν υπάρχουν ούτε τροπολογίες ούτε πρόταση απόρριψης, άρα εγκρίνεται η ε, έκθεση. Και τώρα πάμε στην έκθεση Winkler, αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν οι τροπολογίες που έχουν κατεθεί. Ψηφίζουμε εν σώματι από το 1 μέχρι το 56. Υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται 473 υπέρ. Πάμε στην τροπολογία 7. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. Πάμε στην 11. Ονομαστική ε, ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η 12. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Η 13 ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 28. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 34. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση, αλλά αν τα θέλετε, τέλος πάντων. Για την 28, λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 35. Υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Εντάξει, ηλεκτρονική επαλήθευση. Η 34 ψηφίζουμε παρακαλώ. 34. Ζητήθηκε ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 35. 35. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 36. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 37. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 38. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 38. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 40. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η 41. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. απορρίπτεται. Η 50 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 55 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η 30 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Οι 70 και 111 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 131. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 73, 94 και 114 και 132 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 60 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 74, 95, 115 και 133 είναι ταυτόσιμες σε ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Οι 154 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται. 61 και 22 καταπίπτουν. 75, 96, 116 και 134 είναι ταυτόσιμες ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Οι 76, 97, 117 και 135 είναι ταυτόσιμες. Ονομαστική ψηφορία ψηφισμού. Εγκρίνεται. 77, 98, 118 και 136 ονομαστική ψηφοφορία ψηφι... Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 155. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Κατά ηλεκτρονική επανήλθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Άρθρο 2 η τροπολογία 25 Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες ψηφοφορίες. Πάμε τώρα στο άρθρο 2 το 100 δέλτα. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Υπέρ. Και κοντράρι. Κατά. Αποχές. Δεν έχετε σηκώσει όλοι τα χέρια. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Άρθρο 2. Τροπολογία 138 Δέλτα. Δυνατεύσεω χειρό. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Α, καταπίπτει. Άρθρο 2. Τροπολογία 79, 120 και 139 που είναι ίδιες. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αν ελέγξουμε θέλετε. Ωραία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 101. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογίε 80, 121 και 140 που είναι ταυτόσιμε. Διανατάσσεω τη χειρό, Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογίες 81, 102, 122 και 141 είναι ταυτόσιμες με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Άρθρο 3, τροπολογία 82, 103, 123, 142. Είναι ταυτόσιμες, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 62. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Άρθρο 3, τροπολογία 83, 104, 124, 143. Είναι ταυτόσιμες ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Άρθρο 3. Τροπολογία 63. Διανατάσσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Άρθρο 3. Τροπολογία 64. Διανατάσσεως χειρός υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 84, 105, 125 και 144 είναι ταυτόσιμες με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Άρθρο 4. Παράγραφος 1. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Καταπίπτει. Άρθρο 6. Τροπολογία 32. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται τροπολογίες 86 και 127. Διανατάσσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 146. Διανατάσσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορία. Απορρίφθηκαν. Άρθρο 6. Τροπολογία 33 Δελτά. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ. Να βλέπω τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 6. Τροπολογία 147. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρθρο 6. Τροπολογία 100... Όχι, λάθος. Άρθρο 6, τροπολογία 65, διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ, για να χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 148. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 7. Τροπολογία 66. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 7. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε λοιπόν. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Άρθρο 7. Τροπολογία 42. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται τροπολογίες 87, 108, 128 και 149. Είναι ίδιες. Κάποιος θέλει το λόγο. Ναι, νομίζω ότι για την 66 έχετε κάνει κάποιο λάθος. Πρέπει να ελέγξουμε. Για την 66 με έχει απορριφθεί 66. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι κάνατε λάθος το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Άρθρο 7, τροπολογίες 87, 108, 128 και 149. Με ονομαστική ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Τροπολογίες 129 και 150, πάντα στο άρθρο 7, με ονομαστική ψηφοφορία, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορία. απορρίφθηκαν. 107, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 88. Διανατάσσεως του χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Άρθρο 8. Τροπολογία 68. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 151. Για να τάσω. υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Άρθρο 12. Τροπολογία 152. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ε, μετά το 13, τροπολογίες 89, 109 και 130 είναι ταυτόσιμες με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Άρθρο 15, τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 110. Ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της Απορρίφθηκε. Τροπολογία 58. Διανατάσσεως χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράρτημα 2. 59. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε θέλετε. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη 9. Τροπολογίες 71, 91 και 112 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 57. Τώρα στην ιδεολογική σκέψη 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η τροπολογία 8 και περνάμε στην ατολογική σκέψη 14, τροπολογίες 72 και 92 και 113. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη μετά το 14, τροπολογία 93 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 16, τροπολογία 20, κατά τμήματα. Διανατάστος χειρός, υπέρ του πρώτου τμήματος υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69. Διανατάσσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η πρόταση τροποποιημένη της Επιτροπής τώρα, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Θέλει κάποιος το λόγο. Παρακαλώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, παρακαλώ. Υπάρχουν προβλήματα με το μικρόφωνο από ό,τι φαίνεται. Δοκιμάστε κάποιο άλλο. Δεν λειτουργεί. Μα τι συμβαίνει. Παρακαλώ τις τεχνικές υπηρεσίες να παρέμβουν. Ο Πρόεδρος θέλει το λόγο. Τι έγινε, blackout. Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Περιμένετε, μια στιγμή. Τώρα λειτουργεί. Α, εντάξει. Ωραία. Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, λόγω του αποτελέσματος της ε, ψηφοφορίας ε, που τροποποιήθηκε ουσιαστικά ε, με βάση την ψηφοφορία στην Επιτροπή, με βάση τον κανονισμό 61.2 θέλω μια μικρή διακοπή για να ε, συζητήσω με τον εισηγητή και τους συντονιστές αυτό το νέο αποτέλεσμα. Πέντε λεπτά διακοπή με βάση το άρθρο 61.2. Sì, 5 minuti. questo è possibile? Allora, eh, scusate colleghi. Πρόεδρος, ε, συνάδελφοι, ζητήθηκε η διακοπή της συνεδρίασης για πέντε λεπτά εκ μέρους του Πρόεδρου της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να διακόψουμε για πέντε λεπτά και βεβαίως να καταστεί δυνατόν να υπάρξει αυτή η σύντομη διαβούλευση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Λοιπόν, διακόπτουμε για πέντε λεπτά.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 Ε, Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να καθίσουν. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Presidente Lange. Invito i colleghi a riprendere la loro posizione. Grazie. Presidente Morales. Αν μπορείτε να καθίσετε. Invito i colleghi a riprendere le loro posizioni. Παρακαλώ τους συναδέλφους να καθίσουν. Ξεκινάμε λοιπόν. Υπήρχε αυτό το αίτημα για διακοπή της συνεδρίασης εκ μέρους του Πρόεδρου. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τα συζητήσαμε με τους σκιώδης ηγητές, ε, τον πρόεδρο και τους συντονιστές και τελικά υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά τη συνέχιση των ε, διαβουλεύσεων. Νομίζω όμως επ' αυτού να αποφασίσει η Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν με βάση το άρθρο 61.2 παρακαλώ να διακοπεί η τελική ε, ψηφοφορία και να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Επ' αυτού να ψηφίσουμε. Eh, Πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για αυτό που πρότεινε μόλις τώρα ο πρόεδρος κύριος Λάγκεν. Δηλαδή, το θέμα να αναβληθεί. Υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ να σηκώσει το χέρι. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Votazione chiusa. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η πρόταση. 343 υπέρ, 331 κατά, 9 εποχές. Passiamo ora Περνάμε τώρα στο ψήφισμα το επόμενο ψηφοφορία ε, σχετικά με, την, το κάδμιο πρόταση ψηφίσματος από τέσσερις ομάδες, πολιτικές ομάδες παράγραφος 5 του αρχικού κειμένου ποιος είναι υπέρ παρακαλώ υπέρ, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Στο αρχικό κείμενο, εκτιμώντας F, ψηφίζουμε παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στο ψήφισμα για την ε, εθιλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Επ' αυτού ε, ζήτησε το λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος που είναι αρμόδιος. Παρακαλώ κύριε Επίτροπο. Είμαι αρμόδιος. Well, I'm uh, Εκπροσωπώ πλώς την Κομισιόν, δεν είμαι αρμόδιος. Ε, η Κομισιόν θα ε, ήθελε να σας υπενθυμίσει για τους λόγους αυτούς του κανονισμού που καταργεί, του κανονισμού που καταργεί τον 30, 23-36 ε, της εσωτερικής αγοράς. Η Κομισιόν υιοθέτησε αυτόν τον κανονισμό για την βελτίωση της νομοθεσίας η πράξη αυτή θα άρει τα διοικητικά αχθή για ε, τους εμπορευόμενους ε, χωρίς να επηρεάσει την ε, προστασία ε, των συνόρων θα επιτρέψει την Κομισιόν να συνεχίσει να επιτηρεί την εσωτερική αγορά με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στην συνάντηση της 20 Απριλίου 2015, συνάντησή του, το Συμβούλιο, ε, επιβεβαίωσε ότι δεν, είχε, δεν έχει αντίρρηση για αυτόν τον κανονισμό εξοδοτικής ε, ε, πράξης. Και η Κομισιόν δήλωσε ότι θα επιβεβαιώσει πως θα συνεχίσει να συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία ε, για την παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς με ιδιαίτερη προσοχή στις αγωγές με μηδενικούς δασμούς. Η Κομισιόν καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει ε, την, ε, ε, το αίτημα κατάργησης. Αυτό θα επιτρέψει τη δημοσίευση του κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την θέση του σε εφαρμογή. Πρόκειται για μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ευθυγραμμίσει τη θέση του με τον στόχο μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της απλοποίησης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας κάτι που αποτελεί κοινή ευθύνη ε, Συμβουλίου, Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν επιβεβαιώνει ε, την ε, προσήλωσή της σε μια βελτίωση της νομοθεσίας μέσω του πακέτου βελτίωσης νομοθεσίας που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς ε, κύριε Επίτροπε ψηφίζουμε λοιπόν ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Γεωργίας ε, εκτιμώντας α τροπολογία παριθμών 1 ψηφίζουμε παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται το εκτιμώντας 2 τροπολογία 2 β το 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εκτιμώντα C, τροπολογία 3, με ανάταση χειρός, ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Με ανάταση χειρός, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, επ' αυτού είναι απαραίτητο να ε, ψηφίσει η πλειοψηφία των μελών. Καλύτερα να έχουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζει. La votazione è chiusa. Larga maggioranza, 486 sì. Complimenti. Congedo. Λοιπόν, πάμε στην άδεια μητρότητας. Ψήφισμα, πρόταση ψηφίσματος. Θέλετε κάτι? Παρακαλώ. Θέλετε το λόγο σχετικά με τον κανονισμό? Όχι, διαδικαστικό. Ο κύριος Μπάτεν. Παρακαλώ κύριε Μπάτεν. Είχα την εντύπωση ότι τέτοιες πολιτικές θέσεις δεν επιτρέπονται. Εδώ δεν διαπίστωσα ε, ε, ότι από την άλλη πλευρά του σώματος υπάρχουν διάφορα, διάφορα χαρτιά με συνθήματα. Όμως, αυτό τι σημαίνει, ότι πολιτικής φύσης πόστερ μπορούν να κυκλοφορούν εδώ στην Ολομέλεια. Τότε εντάξει, και εμείς. Διακόπτει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπάτεν συνεχίζει. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορούμε για να το κάνουμε και εμείς. Πρόεδρος. Κοιτάξτε κύριε Μπάτεν, Θέλω να σας πω ότι αυτό που κάνετε τώρα δεν ε, προβλέπεται στον κανονισμό. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε όπως και το να συζητήσουμε το θέμα των ε, σημαίων ε, κρατών στα έδρανα των προβλεπτών. Αυτό κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε. Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Μιλάμε και ψηφίζουμε για την πρόταση ψηφίσματος άδεια μητρότητα σε πρώτη παράγραφο σε δύο τμήματα με ανατεσχυρός υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ανατεσχυρός υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση, ψηφίζουμε. Παράγραφος 4. 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 3 ψηφίζουμε σε δύο τμήματα δυνατά χειρός υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα τώρα πάντα δυνατά χειρός υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήτευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία υπέρ 1. Δυνατά σε χειρός υπέρ. Κατά επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στο εκτιμώντας F υπέρ, κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε, ε, ε, ψηφίζουμε για το σύνολο του, ε, της πρώτης ψηφίσματος με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Πρόταση ψηφίσματος από 7 πολιτικές ομάδες. Τροπολογία υπαριθμών 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Διανατάσεως χειρός. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντα εκτιμώντας ε, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του δυνατά χειρός υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πολύ ωραία και συγχαρητήρια. Και τώρα Ψηφίζουμε για την πρόταση ψηφίσματος επιδημίας ξυλέλαφα στην ένα βακτήριο που προσβάλλει τα ελαιόδαντρα. Πρόταση ψηφίσματος από δύο πολιτικές ομάδες. Ψηφίζουμε παρακαλώ με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. απορρίπτεται. Κατόπιν τούτου ψηφίζουμε για το κοινό ε, ψήφισμα, κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τέσσερις πολιτικές ομάδες, παράγραφος 1 του αρχικού κειμένου, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3 του αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα, διανατάσσεως της χειρός, πρώτο τμήμα παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, δυνατάσσεως χειρός, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, πάντα διανατάσεις χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 με ονομαστική ψηφοφορία, ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Στη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 19. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 16, ε, δυνατός χειρός, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Η 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 18. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 20. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική παλήθευση. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτηκε. Τροπολογία 22. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η τροπολογία 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές επαλήθευση ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ή οι τροπολογίες, οι 3 και οι 12 που είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Η 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 13. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 5 και η 14 είναι ταυτόσιμες. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η έξι, Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η επτά, Με ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε ψηφο... Ε, ε, ψηφίζουμε, με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε τώρα. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε τώρα για το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται το ψήφισμα.